η ψηφοφορία αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Επόμενο σημείο, η έκθεση της κυρίας Φώστερ για την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ε, τον λόγο έχει η συγγήτρια για 4 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το 2012 είναι κέντρο ε, χρονιά σημαντική για το έργο των του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Μετά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσα πολλά από τα θέματα Τη δική μου ε, ε, έκθεση ιδιαίτερης πρωτοβουλία που υποστηρίξαν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή ε, Μεταφορών και Τουρισμού τον Ιούλιο. Η εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού έχει ξεπεράσει πολλές περιορισμού και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλέ δυσκολίε. Η ευρωπαϊκή κυκλοφορία συνεχίζει να αυξάνεται, πράγμα που είναι καλό για την ανάπτυξη, αλλά δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα στα περισσότερα κράτη-μέλη. Πρέπει να αισθανθούμε περισσότερο την αίσθηση του επίγοντο για να αντιμετωπίσουμε τους επιχειρησιακούς κινδύνους με τους αυξανόμενες ροές κυκλοφορίας. Τα ωφέλη μιας πλήρους και έγκαιρης εφαρμογής του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού είναι σαφή και δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Η μελέτη της κοινή επιχείρησης ΕΖΑΡ δείχνει ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 300.000 θέσει εργασίας, θα γίνουν εξοικονομήσεις πάνω από 50.000 τόνων ε, διοξείδου του άνθρακο και θα γίνει πιο αποτελεσματική η ενέργεια κυκλοφορία, θα μειωθεί το κόστος για τον καναλωτή και Βεβαίω, θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στο παγκόσμια αγορά για να διατηρήσουμε το μερίδιό μα. Αυτό είναι πολύ καλή επιχειρηματική πρακτική και μόνο και μόνο για αυτού του λόγου είναι σαφέ ότι το να γίνει ο ευρωπαϊκός εναέριο χώρος όσο το πιο αποτελεσματικό, είναι καλό για τι θέσει εργασία και το περιβάλλον. σε μια περιοχή που πολλές, ε, περίοδο που πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε πηγαίνουν προ την ύφωση τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικά. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα θα είναι αντιληπτά σε όλα τα κράτη-μέλη και θα καλύψουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών, των αεροπορικών εταιριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τομεί όπω ο τουρισμό. Είμαι πεπισμένη κύριε Πρόεδρε ότι οι θέσει εργασία που θα δημιουργηθούν θα είναι υψηλών δεξιοτήτων και υψηλών αμοιβών. Το ΣΕΖΑΡ θέλει οι ελεγκτέ ενεργείου κυκλοφορία να γίνουν ένα πιο ευκίνητο εργατικό δυναμικό και να μπορούν να πουλάνε τι δεξιότητέ του ευρύτατα και να συνεισφέρουν σε ένα πιο ισχυρό και καινοτόμο τομέα κατάλληλο για τον 21ο αιώνα. Μια από τι βασικέ προκλήσει είναι ο, ο των Ευρωπαίων ε, του ευρωπαϊκού ε, ουρανού. Η προόδος είναι ε, βραδία και απαράδεκτη. Πρέπει να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στα κράτη-μέλη, γιατί είναι αυτά τα ίδια κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει για το έργο αυτό εδώ και πάνω από 10 χρόνια, όταν για πρώτη φορά φέραμε αυτή την νομοθεσία. Και επιπλέον, οι χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Εμείς στην Ευρώπη είμαστε ηγέτες στην ανάπτυξη τεχνολογίας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δικές μας εταιρείες θα υποφεληθούν από αυτήν. Είναι ζωτική σημασία να συνεργαστούμε στενά με τις γειτονικές χώρες και με το στρατιωτικό τομέα για να εξασφαλίσουμε ότι τα συστήματα που αναπτύσσουμε ε, θα έχουν διαλειτουργικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι, οι, οι, οικονομικές επενδύσεις έρευνα και ανάπτυξη για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό είναι σημαντικές και πλέον τώρα πρέπει να τεθούν τα απαραίτητα τα μέτρα για να ε, ε, αποκομίσουμε τα ωφέλη αυτών των επενδύσεων. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι κουράστηκα να ακούω τα προβλήματα και για το τι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, όταν στην ουσία είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις. Επίσης ανταγωνιζόμαστε με τις ε, αναδυόμενες αγορές Ασίας, Νότιας Αμερικής και Μέση Ανατολής. Και είτε θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, είτε θα υποστούμε τις συνέπειες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να σταματήσουν την κολυσιεργία και να προχωρήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη στήριξη του Κοινοβουλίου για να επιβάλλει κυρώσει στα κράτη-μέλη που δεν ε, συμμορφώνονται. Με την ευκαιρία αυτή, ο Επίτροπος Κάλλας, που δεν βρίσκεται σήμερα εδώ, έχετε την πλήρη ε, υποστήριξή μου και ελπίζω να προχωρήσετε με πλήρη ισχύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Περνάμε στη διαδικασία και τη Το λόγο έχει η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ενέργειο χώρος πρέπει να γίνει πραγματικότητα και θα πρέπει να τον χρησιμοποιούμε με τη μέγιστη ασφάλεια. Αυτό θα ευεργετήσει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, αλλά και το περιβάλλον. Επιπλέον έχουμε, θα έχουμε ένα πιο αηφόρο σύστημα αεροπλοείας. Οι πρόοδοι που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα πρέπει να υποστηριχθούν και να συνεχιστούν. Εμείς χρειαζόμαστε αεροπορικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας κυρίως σήμερα όπου η, κυκλο, ε, ενέργεια κυκλοφορία αυξάνεται σε, ε, συνεχώς. Χρειαζόμαστε ομοιογένεια σε όλα τα κράτη-μέλη και χρειάζεται συνεργασία και σύμπραξη. Ευχαριστώ κύριος Δανέλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τον Απρίλιο του 2010, όταν ταλαιπωρήθηκαν περισσότεροι από 100.000 επιβάτες από την έκρηξη του Ισλανδικού ηφαιστείου, τα κράτη μέλη έσπευσαν να διακηρύξουν πως ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός δεν μπορούσε να επιδειχθεί καθυστερήσεων. η ευρώπη χρειάστηκε και δεν είχε την ευελιξία ενός κοινού ενέργειου χώρου. δυόμιση χρόνια μετά βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο όπου η άμεση ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού φαντάζει μάλλον ουτοπική ενώ καθυστερεί ακόμη και η τυπική θέσπιση των ΦΑΜΣ που από μόνη της εξάλλου δεν εγγυάται βελτίωση των επιδόσεων των αερομεταφορών. αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι να υπερισχύσει η πολιτική βούληση της γραφειοκρατίας και των συμφερόντων της ακινησίας να καμφθούν οι εθνικοί εγωισμοί και γι' αυτό ειδικά σήμερα ας μην παραβλέπουμε τη βαρύτητα και του συμβολισμού. ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι ένα τεχνικό έργο με γνωστά ωφέλη αναφέρθηκαν ήδη αλλά είναι ταυτόχρονα ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αυτό ας το θυμόμαστε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Δανέλη. Ολθεί ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός ευθύς εξ αρχής ήταν, ε, είχε συσχετιστεί με την απελευθέρωση των μεταφορών. Ο βασικός στόχος εδώ δεν ήταν ε, να αναπτυχθεί ο τομέας προς όφελος των επιβατών, αλλά να μπορέσει ο ευρωπαϊκός ουρανός να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες των πολυεθνικών εταιριών και των αεροπορικών εταιριών το συμφέροντα των ε, επιβατών υπόκεινται 100% στα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών και αυτό στοιχίζει ε, θέσει εργασίας και στοιχίζει στο περιβάλλον όπως επίσης στοιχίζει και στις δημόσιες ε, κρατικές αεροπορικές εταιρείες και άλλες εταιρείες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ό,τι συνέβη και τι θα πρέπει να συμβεί. Χρειάζεται καλύτερη χρήση του χώρου και κάθε κράτος μέλος να κρατήσει ανοιχτό τον εναέριο χώρο του. Αυτό είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση των οικονομιών των χωρών μας και για την οικονομία και για την άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύμφωνο 100% με την κυρία Φώστερο όταν λέει ότι έχουμε τεράστια καθυστέρηση για τη δράση, στη δράση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις. Πράγματι, στην Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την καινοτόμο τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να μας βοηθήσει και με μεγάλα οικονομικά έσοδα. Με αυτή την επανοργάνωση θα έχουμε 419 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδος, 328.000 θέσεις εργασίας και ένα σωρό ε, τόνοι διοξιδίου το άνθρακος λιγότερο. Πρέπει να σκεφτούμε και στην κατάρτιση του προσωπικού, διότι στην, στην Ανατολική Κεντρική Ευρώπη είμαστε πολύ πιο κάτω από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετανάστευση από αυτές τις χώρες προς άλλες. Ευχαριστώ κύριε Τσικάου. Ο, ο ενιαίος ε, ευρωπαϊκός ουρανός απαιτεί ενίσχυση των όρων ασφάλειας και αυτή η ασφάλεια μας ε, τονίζει την ανάγκη προγραμμάτων όπως ο Γαλιλαίος και την ανάγκη ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ουρανού. Σύμφωνα με την Κομισιόν η εισαγωγή του ΣΕΖΑΡ θα οδηγήσει θα, θα βοηθήσει ιδιαίτερα τους επιβαδές, θα μειώσει 10% την διάρκεια των πτήσεων, θα μειώσει τα εισιτήρια, θα μειώσει τις καθυστερήσεις. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό υπό όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ακόμη και τα περιφερειακά. Και αυτό για να αποσυμφορηθούν τα δίχτυα και η εναέρια κυκλοφορία. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Τελειώνουμε με τον κύριο Μικολάτσικ, το Κατστιάη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο, ο ευρωπαϊκός χώρος ε, της ε, ενέργειας κυκλοφορίας είναι ο πιο φορτωμένος στον κόσμο και, αυτό θα, και θα πρέπει ο, το βάρος αυτό να διπλασιαστεί μέχρι το 2020. Άρα θα πρέπει το, ε, το σύστημα αυτό του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού να εφαρμοστεί, να εγκατασταθεί γέρος έτσι ώστε ε, να επηρεαστούν θετικά ε, τα 27 κράτη-μέλη και στο ΑΕΠ τους και στις θέσεις εργασίας με τη δημιουργία 300.000 θέσεων εργασίας με την εξοικονόμηση των 50 εκατομμυρίων τόνων ε, διοξιδίου του άνθρακος. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να παλέψουμε για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ΘΙΑΗ. Τον λόγο έχει ο Επίτροπος ο κ. Πίμπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η έκθεση για την εφαρμογή του Νέα Ευρωπαϊκού Ουρανού έρχεται σε μια στιγμή κρίσιμη. Έρχονται Σύντομα πάρα πολλές προθεσμίες. Το 2012 είναι έτος κρίσιμο. Έχουμε τέσσερα κρίσιμα παραδοτέα μεταξύ των οποίων εννέα μπλοκ εναερίου χώρου που θα πρέπει να είναι επιχειρησιακά μέχρι το Δεκέμβριο. Οπότε καλωσορίζουμε την έκθεση και ευχαριστούμε την Επιτροπή Μεταφορών και την κυρία Φώστερ. Η εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου στην Λεμεσό προσφάτως. Το βασικό συμπέρασμα των συζητήσεων είναι πώ η πρόοδο είναι αργή και τα πλέον δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει ακόμα μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και υπάρχει μια κατακαιρματισμένη προσέγγιση που βασίζεται σε ε, ε, ε, στα εθνικά όρια. Κάτι το οποίο προσθέτει κάθε χρόνο 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο κόστος αεροναυτιλίας. Υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα πρόβλημα χρόνου. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα και να προχωρήσουμε με την εφαρμογή. Ένας από τους λόγους για αυτή την κατάσταση φαίνεται πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν πρόσφατα απέθυνε επιστολή στους Υπουργούς Μεταφορών υπενθυμίζοντάς τους τις ε, υποχρεώσεις τους για να δράσουν γρήγορα και εγκαίρως. Θα αυξήσει η Κομισιόν τις προσπάθειές της για να υπάρξει μια έγκαιρη και γρήγορη εφαρμογή. Εάν υπάρξει ανάγκη, η Κομισιόν θα προσφύγει κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται. Δεύτερον παρά το ότι έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την συμμόρφωση και προς την υλοποίηση αποτελεσμάτων. Συμφωνώ μαζί σας πως ο πυλώνας της απόδοσης πρέπει να ενισχυθεί και να έχουμε συγκεκριμένα επιχειρησιακά ωφέλη τα οποία θα υπάρξουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των λειτουργικών μπλοκ αερίου χώρου. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αξιολογεί μέτρα για να επιταχύνει την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού ουρανού για να μπορέσουν να απελευθερωθούν τα θετικά και συμφωνεί η Κομισιόν να δίνει αναφορά στο Κοινοβούλιο ξεκινώντας από το 2013 όσον αφορά την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού καθώς και όσον αφορά τη στρατηγική μας για μια πιο αποφασιστική εφαρμογή. Οι αρχές της υφιστάμενης νομοσίας εξακολουθούν να ισχύουν. Δεν χρειάζεται να ξανασχεδιάσουμε τίποτα από την αρχή. Πρέπει απλά να κάνουμε κάποιε αλλαγέ για λόγους ταχύτητα και αποτελεσμάτων. Πρέπει να απλοποιήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε την νομοθεσία. Επίσης μπορώ να σας ενημερώσω πως ήδη επεξεργαζόμαστε νέες προτάσεις για να επιταχύνουμε την εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Να συμπληρώσουμε κάποιες ατελείς πρωτοβουλίες και να ενισχύσουμε την εξτάμενη νομοθεσία πρόθεσή μας είναι οι προτάσεις αυτές να δημοσιευτούν την άνοιξη του 2013. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και αυτή η ψηφοφορία αύριο στις 6 ώρα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη έκθεση Μπαχ